Bueno, continuamos si les parece y comenzamos con las votaciones. Να συνεχίσουμε και να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Έχουμε λίγο καθυστερήσει. Έχετε τις ε, κάρτες Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ψηφίζουμε το σημείο 10. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Πρώτα απ' όλα να ψηφίσουμε από κοινού τα σημεία 10, 11 και 12. υπάρχει κάποια κάρτα που δεν λειτουργεί. Τι γίνεται. Λοιπόν, παρακαλώ λίγη ησυχία για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε το σημείο 10, το σημείο 11 και το σημείο 12 από κοινού. Απόλυτη πλειοψηφία απαιτείται. Μάλλον πρέπει να σας τα εξηγήσω. Δυνάμει του άρθρου 70 αναθεωρήθηκε πρόσφατα. Ε, πρόκειται για τη τρομολόγηση διοργανικών διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, παρακαλώ λίγη ησυχία. Αν μιλάτε όλοι ταυτόχρονα, αδύνατον να καταλάβετε και τι σας λέω και γι' αυτό αμφιβάλλετε. Λοιπόν, αν με επιτρέπετε, ακούστε με, για να είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Για να μπορέσουν λοιπόν να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις, κομισιών πρέπει να υιοθετήσει μια επίσημη συμφωνία με απόλυτη πλειοψηφία των μελών. Η Επιτροπή μας συγκεκριμένα για την τελή διαπραγμάτευση και τη σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας. Έχετε το έγγραφο, το σχετικό και το, τους τίτλους τους ξέρετε, τους ηγητές τους ξέρετε, την διαπραγματευτική ομάδα την ξέρετε, τη μέρα που εγκρίθηκε την ξέρετε. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να ψηφίσουμε την απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων, δύο οργανικών διαπραγματεύσεων, για τις τρεις διαδικασίες τις οποίες σας ανέγνωσα, δηλαδή τα σημεία 10, 11 και 12. Συμφωνείτε, υπάρχει κάποια αμφιβολία. Ωραία. Όλα είναι ξεκάθαρα. Άρα θέτω σε ψηφοφορία τα τρία σημεία, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίθηκε. 19 ψήφοι υπέρ, μία κατά, μία αποχή. Απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, όπως είπαμε. Στον κύριο Ρεβελίν δεν λειτουργήσε η κάρτα. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως δεν θα άλλαζε το τελικό αποτέλεσμα. Αν συμφωνείτε μπορούμε να συνεχίσουμε. Και περνάμε στο σημείο 13. την έκθεση του κυρίου Κούν. Τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου στο σκάγκερα και τροποποίηση των κανονισμών αυτών. Περνάμε γρήγορα αν ε, δεν έχετε αντίρρηση. Τροπολογία 10 Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Με μία ψηφοδιαφορά. 11 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 12 τροπολογία άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 55 τροπολογία άρχεται. Ψηφοφορία. Πέρασε. Εντάξει, την ξαναρχίζω, την ξανακλίνω. Εγκρίνεται. 13 τροπολογία άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 14 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε εγκρίνεται. 15 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Όχι. Ξαναρχίζουμε. Τώρα κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα. 56 υπέρ. 56. Ψηφίζουμε έτσι. Απορρίφθηκε. Τώρα 19. Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. 19 Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 63. Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Λάθος. 21 λοιπόν. 21 τροπολογία. Άρχεται. Ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία που πάμε. 22. 22. του ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 70. 70, 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και τώρα, συμβιβαστική 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, η πρώτη και τρίτη παράγραφος. Α, έχει πέσει, καταπέσει το δεύτερο τμήμα, Ψηφίζουμε μόνο το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 75. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. 76 έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. 24 έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. 77 έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5α. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε την 5β και πάμε στην 84. Όχι. Πάμε στη συμβαστική 6. Έναρξη ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Έναρξη ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 35 τροπολογία. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 103. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 105, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 106, έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. 38. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμπεριβαστική 8. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. 114. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Για να δούμε τι έγινε με την 37 πρώτα όμως. Λοιπόν, τροπολογία 2. Έναξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Έναξη ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. Σαράντα plus. 46. τροπολογία. Έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. Επτά Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 8 τροπολογία τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 49. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την τροποποιημένη νομοθετική πρόταση έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας εγκρίνεται. Εγκρίνεται λοιπόν τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, έναρξη ψηφοφορία. πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Κούν. Μία αποχή μόνο είχαμε. Επόμενο θέμα. Ψηφοφορίζουμε την αλλαγή του κανονισμού 812 για τα παρεμπίπτωτα το κοιτοειδών κατά την αλληλεία και την τοποποίηση του κανονισμού 88 του 98 με τον κύριο Ρομέβα. Τροπολογία 5. Άρχεται. Πέρας. Επαναλαμβάνουμε για την τροπολογία 5. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Άρχεται, συγγνώμη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροποποιημένη η νομοθετική πρόταση όπως, ε, όπως έγινε. Άρχεται. πέρα Εγκρίνεται. Και το ψήφισμα, το νομοθετικό ψήφισμα άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Ρωμέβα. Επόμενο. Απαλλαγή 2011. Κοινωνική υπηρεσία ελέγχου της Αλίας. Ε, απαλλαγή 2011. Γενικός προϋπολογισμός Ένωσης τμήμα 3 με εισηγητή τον κύριο Τόρφαλτς. Τροπολογία 1. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Άρχεται. Περαιούται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Άρχεται. Περαιούται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται. Περαιούται. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης. Άρχεται. Περαιούται. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Προς τον κύριο Τόρβαντ. Σημείο 16. Έγκριση της απαλλαγής 2011 την κοινωνική υπηρεσία ελέγχου αλίες. Με συντάκτη γνωμοδότηση του κύριο Σαλαβράκο. Δύο τροπολογίες. Ε, τροπολογία 1. Άρχεται. Περαιούται. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 άρχεται. Περαιούται. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης. Άρχεται. Περαιούται. Εγκρίνεται με μία αποχή. Συγχαρητήρια. Κύριε Σελαβράκο, με αυτό κλείνουμε τις ψηφοφορίες. Προχωρούμε στη συζήτηση. Προτείνω, αν συμφωνεί η κυρία Ντότς, που είναι η συγγήτρια των δύο θεμάτων, 5 και 6, μαζί μπορούμε να τα δούμε νομίζω αν συμφωνείτε. Είναι πιο γρήγορο. Συμφωνείτε κυρία Ντότς. Άρα συζητούμε το σημείο και το σημείο 6. Ακούσαμε την παρουσίαση της Επιτροπής, είχαμε και δύο ανταλλαγές απόψεων για την πρόταση. Προτείνω να εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης της συγγήτριας μαζί και για τις δύο εκθέσεις, με ενιαία παρέμβαση. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Εντάξει. Κύριε Ντότς, έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, εμείς ε, προτιμάμε να υπάρξει μία ε, αρχική συζήτηση ε, σχετικά με την έκθεση αυτή και μετά να ακολουθήσει μια πιο ουσιαστική συζήτηση για τη δεύτερη έκθεση που κατά την άποψή μας ε, περιλαμβάνει πολλές ε, περισσότερες λεπτομέρειες και είναι και πρακτικής φύσεως η έκθεση αυτή. Και οι λόγοι θα καταστούν ε, σαφείς καθώς θα προσπαθήσω να κάνω και τον διαχωρισμό ανάμεσα στις δύο εκθέσεις. Όσον αφορά την πρώτη έκθεση, θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία του Συμβουλίου ε, για το ότι μας βοήθησε σε αυτές τις εκθέσεις. Βρίσκομαι σε μία μοναδική θέση, δηλαδή παρουσιάζω δύο ε, σχέδια εκθέσεων. Ο πρώτος ε, αφορά την διαδικασία προσαρμογής στη συνθήκη της Λισαβόνας και θα θυμάστε τι έχει προηγηθεί. Η δεύτερη έκθεση τροποποιεί τον ίδιο κανονισμό με έναν πρακτικό και ουσιαστικό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα, προτιμούσα να εστιάσω στη διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο εκθέσεις, ε, κυρίως σε σχέση με τα σχόλια της Κομισιόν σήμερα το πρωί. Ε, στη... Σήμερα θα ήθελα επίσης να πω το εξής. Υπάρχουν και επικαλύψεις σε όλο αυτό το θέμα των μακροχρόνιων προγραμμάτων διαχείρισης. Και αυτή είναι μια συζήτηση που νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε, μια συζήτηση η οποία φαντάζομαι ότι θα διευκρινίσει ορισμένα θέματα, αλλά και απόψεις της Επιτροπής σχετικά με το ευρύτερο θέμα. Οι αποφάσεις λοιπόν που ελήφθησαν από τους Υπουργούς Αλίας στις 18 Δεκεμβρίου του 2012 μπορούν ε, να προσφέρουν την ευθυγράμμιση των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων για το γάδο και επίσης ε, μπορούμε με τον τρόπο αυτό να αποκτήσουμε και λίγο χρόνο για να συνεργαστούμε με την Ιρλανδική Προεδρία έτσι ώστε να ζητήσουμε λύσεις ε, στα προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι αξίζει τον κόπο να δούμε λιγάκι το χρονοδιάγραμμα που οδήγησε σε αυτή την απόφαση ο κανονισμός 1342 του 2008 που πρόβλεπε για πρώτη ε, φορά ε, μακροχρόνιο ε, προγραμματισμό για το γάδο. Αυτό αποφασίστηκε το 8 και αργότερα τέθησε ισχύ. Το πρόγραμμα λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να ε, εμπλουτιστούν τα αποθέματα του ΓΑΝΤΟΥ και προβλεπόταν ότι θα υπάρξει αναθεώρηση μετά από τρία χρόνια εφαρμογή. Έγινε λοιπόν αναθεώρηση από την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Ελίας που δημοσίευσε τα ε, σχόλιά της ε, στις θάλασσες που έκανε τις έρευνες στην Κοπενχάγη ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αυτά και έγινε αποδεκτό ότι μόνο μετά από τρία χρόνια εφαρμογής του προγράμματος ήταν πάρα πολύ νωρίς ε, να ε, συμπεριληφθούν ε, τα προγράμματα σε τελική φάση. Κατέληξε όμως ότι το πρόγραμμα αυτό δεν προβλέπει σχόλια για την θνησιμότητα των ε, ψαριών και σε πολλές ε, περιοχές ε, δεν προβαίνει σε απολογισμό. Αυτό θα ακολουθήσει διότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ενέργειες των εμπλεκομένων. Εξάλλου, θεωρητικά, η υποστήριξη αυτού του προγράμματος οδηγεί στην αποδοχή των ευθυνών και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Έτσι λοιπόν καταλήγω στο ότι ε, είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα νέο σχέδιο και αυτό γίνεται αποδεκτό από την Επιστημονική Επιτροπή. Η Επιτροπή χρειάστηκε άλλους 14 ε, μήνες για να δημοσιεύσει τις ε, αλλαγές που προτείνει στο πρόγραμμα αυτό. Αυτά συνέβησαν το Σεπτέμβρη του 2012. Βεβαίω είναι πήγον να λυθούν κάποια προβλήματα που σχετίζονταν με το πρόγραμμα και έτσι λοιπόν η Κυπριακή Προεδρία προσπάθησε να λύσει κάποια θέματα που είχαν σχέση με τα ανώτατα επιτρεπτά αλλιεύματα γάδου. Η πρόταση της ε, Προεδρίας ήταν να αντιγράψει τα άρθρα 9 και 12 από την πρόταση της Κομισιόν του Σεπτεμβρίου του 2012. Ε, επίσης, ε, το Συμβούλιο αναφέρθηκε στα άρθρα 43.2 και 43.3 της Συνθήκης Λισαβόνας. Εκεί αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει κάποια αρμοδιότητα και Συγγνώμη, ε, διαβάζετε με πολύ μεγάλη ταχύτητα κυρία Ντότζ και το Κοινοβούλιο νομίζουμε ότι απέρριψε λοιπόν ε, αυτές τις προτάσεις ε, και αυτά παραπέμπτηκαν για δικαστική γνωμοδότηση. Υπάρχει τώρα το επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης, ε, το οποίο νομίζω ότι έχει περισσότερη ουσία, γιατί πρέπει να συζητήσουμε τις ε, τροπολογίες που πρέπει να κατατεθούν. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει εδώ να συζητήσουμε για το πού κατά την άποψή μας κατευθύνεται το όλο θέμα. Εγώ λοιπόν δεν τάσομαι υπέρ της ε, ε, επιλογής ε, της δικαστικής οδού αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο προτιμούν βέβαια να καταφύγουν στο δικαστήριο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτό παραπέμπεται στις καλένδες, ε, θα λέγαμε απλά, και σημαίνει επίσης ότι το Συμβούλιο δεν βλέπει κανένα απολύτως λόγο να μετακινηθεί από τη θέση του. Γι' αυτό λοιπόν ε, καλώ την Επιτροπή να μην πέσει σε αυτή την παγίδα και η επιλογή της ε, Δικαστική οδού να παραμείνει ανοιχτή για εν χρόνο, για επιλογή εν ευθέτω χρόνο. Θα έλεγα επίσης ότι αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να υπάρξει μία πρόταση από την Ιρλανδική Προεδρία, από κοινού με την πρόταση της Επιτροπής, ε, τη σημερινή πρόταση και έτσι μπορεί να υπάρξει συνεργασία για αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση προσαρμογής, για να προχωρήσει η έκθεση αυτής της Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις απόψεις της ε, δικής μας Επιτροπής για το θέμα αυτό. Όσον αφορά τις ε, τροπολογίες, εγώ προσπάθησα να ενισχύσω τη θέση του Κοινοβουλίου και της ε, επιστημονικής ε, γνωμοδότησης, αυτά να τα εντάξω στη διαδικασία ευθυγράμμισης και βεβαίως σας είπα ότι με μεγάλη μου χαρά να ακούσω και τις ε, δικές σας απόψεις για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστούμε κυρία Ντότζ. Κύριος Βαλένσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω για το σημείο 5. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανείς με τις τροπολογίες της και επιπλέον είναι θετικό το ότι η κυρία Ντότσε ε, επέκτηνε, επεξέτεινε την ανάγκη συμβουλευτικής ε, περιφερειακών περιφερειακών ε, οργανισμών. Νομίζω ότι πρέπει η Ένωση να ακούει τις απόψεις των περιφερειακών δομών πριν λάβει φάσεις ε, για νέες τιμές και όγκους. Την ευχαριστώ λοιπόν για το σημείο 6 τώρα. Στην προηγούμενη συνάντηση συμφωνήσαμε όλοι ότι ο κανονισμός αυτός είναι άλλο ένα παράδειγμα μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου που δεν σχετίζεται με την πραγματικότητα και κατά συνέπεια δεν έδωσε τα αποτελέσματα, δεν βελτίωσε δηλαδή την κατάσταση των αποθεμάτων γάδου. Η συγγήτρια υπογράμμισε εκ νέου την ανάγκη επιστημονικής συμβουλευτικής με νέες τροπολογίες που υποστηρίζουμε. Η τροπολογία 4 διευκρινίζει την ανάγκη να τηρούνται όλα τα κριτήρια και το ίδιο αφορά την παράγραφο 6 που, που απλοποιεί τις διοικητικές διαδικασίες. Τις υποστηρίζω, διότι είναι λογικές. Ωστόσο, δεν υπάρχει σωστή διατύπωση ακόμα για το άρθρο 11, ιδίω το σημείο Γ. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής στην τροπολογία 5, που την εξετάζουν και οι δικοί μου ειδικοί και ελπίζω να έχω κάποια αποτελέσματα σήμερα ήδη. Θα συνεχίσω να υποβάλω τροπολογίες βάσει των δικών μου παρατηρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει για την έκθεση. Είχαμε κάποιες δυσκολίες ε, χρονικού χαρακτήρα γιατί τα Χριστούγεννα του Συμβούλου αφαίρεσε ορισμένες σημαντικές διατάξεις από τον κανονισμό για τα ΤΑΚ. Νομίζω ότι σωστά έκανε η εισηγήτρια εξετάζοντας τις συνέπειες της απόφασης του Συμβουλίου και εμένοντας στη θέση ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να μετέχει στις διαδικασίες αυτές. Υποστηρίζω λοιπόν τις τροπολογίες 2 και 3 για τις διαδικασίες ε, σχετικά με το ΤΑΚ. Χρειάζεται ευελιξία για τις επιστημονικές θέσεις και τον τρόπο διαμόρφωσης των ποσοστώσεων. Πιστεύω επίσης ότι υπάρχουν και άλλες μέθοδοι για να πετύχουμε κάτι τέτοιο και να μειώσουμε τις ποσοστώσεις και για τα αποθέματα για τα οποία υπάρχει τεκμηρίωση και για εκείνα όπου δεν υπάρχει. Επίσης υποστηρίζω στο τροπολογίες 8 και 9. Θετικά είμαι τέλο πάντων ε, διακείμενος. ευθυγραμμίζονται με τις δανεικές διατάξεις για, τα μεταβιβάσιμα, για τις μεταβιβάσιμες ποσοστώσεις. Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα προβλήματα, μακροπρόθεσμα προβλήματα που σχετίζονται με τις ποσοστώσεις και περιμένω να δω τις, τα προγράμματα της Επιτροπής για τα μεικτά αλλιεύματα και θα έπρεπε να έχουμε μια διευκρίνηση για την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στο πλαίσιο αυτό, όταν βλέπουμε τα μακροπρόθεσμα σχέδια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο κύριο Στίβενσον. Ευχαριστώ. Αυτό που έκανε το Συμβούλιο το Δεκέμβριο ήταν απαράδεκτο. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να φωνάζουμε στο Συμβούλιο όπως κάνουμε το πρωί. Είπαμε τι είχαμε να πούμε και αν συνεχίζουμε να φωνάζουμε ε, χάνουμε το δίκιο μας. Εάν τους πάμε, το είπε και η κυρία στο δικαστήριο, είναι ο καλύτερος τρόπος να, να, να, μείνουν στις θέσεις τους και να μην γίνει τίποτα. Άκουσα την Επίτροπο το πρωί να λέει ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε με δύο στόχους. Πρώτον, να επιδιώκουμε ένα συμβιβασμό, να δούμε το συμβασμό που πρότεινε η Επίτροπο και νομίζω ότι είναι ευκαιρία και να συζητήσουμε την ιδέα αυτή. Ταυτόχρονα δε, να πάμε και στο δικαστήριο. Και πάλι ωστόσο δεν θα υπάρχουν συζητήσει στο Συμβούλιο για οποιοδήποτε συμβιβασμό αν εμείς πάμε στο δικαστήριο. Θα χρησιμοποιήσουν το επιχείρημα αυτό σαν την κάρτα αποφυλάκησης, αν θέλετε, που δεν θα έχει εναλλακτική λύση για αυτούς. Νομίζω ότι, όπως είπε και η κυρία Δαμανάκη, υπάρχει μια αντίστοιχη, παρόμοια, σχεδόν ίδια περίπτωση, που έχει πάει στο δικαστήριο η Επιτροπή και τρέχει. Ας δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση και ας συζητούμε ταυτόχρονα για πιθανούς συμβιβασμούς. Καταλαβαίνω ότι μετά τη το γεύμα που είχε πριν από δύο εβδομάδες ο κύριος Κόβανη, ο, προεδρεύων, ο Προεδρεύων, οι Γάλλοι που είχαν την πιο σκληρή θέση επανήλθαν με μία επιστολή προτείνοντας, λέγοντας μάλλον ότι δεν θέλουν να υπάρξει μία σκληρή μηχανοποιημένη προσέγγιση καθορισμού τάκ και ποσοστώσεων, αλλά θα μπορούσαν ίσως να συζητήσουν για άλλα θέματα. Αυτό ήταν ε, η πρώτη αχτίδα φωτός που δείχνει ότι κάπως μαλακώνει η γαλλική θέση. Μπορεί να μην είστε τόσο αισιόδοξοι, βλέπω ότι νεύετε αρνητικά, αλλά τέλος πάντων. Θα μπορούσαμε αυτό να το δούμε ως ένα πιθανό, μια πιθανή ακτίδα φωτός στην άκρη του τούνελ. Τέλος, η συμβιβαστική λύση που πρότεινε σήμερα το πρωί η Επίτροπο ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει πριν από ένα χρόνο στην Επιτροπή μα. Όπου εμεί θα, λέγαμε, θα δίναμε το OK στην αρχική διαμόρφωση του πλαισίου του πολιετού προγράμματο, κατόπιν ωστόσο το αφήνουμε στο Συμβούλιο να εφαρμόσει τυχόν αναθεωρήσει. Είπα το πρωί στην κυρία Δαμανάκη, το επαναλαμβάνω τώρα. Αυτό είναι λογικό. Αν μπούμε στις διαδικασίες αναθεώρησης ξανά και ξανά, η διαδικασία συναπόφασης καθυστερεί τα πάντα. Και εμένα μ' αρέσει να μετέχει το Κοινοβούλιο στην αναθεώρηση, στην τακτική αναθεώρηση των πολιετών προγραμμάτων. Δεν είναι πρακτικό, δεν είναι λογικό. Αν λοιπόν έχουμε απόλυτο λέγειν στη διαμόρφωση του πλαισίου για τα πολιετή προγράμματα, τούτο είναι μια συμβιβαστική λύση θετική που θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη. Και αν η Επιτροπή δουλεύει μαζί μας ως σύμμαχος για να διευκολύνει τον συμβιβασμό, θα, βρούμε, θα δούμε το τέλος αυτού του μακρού δρόμου. Ας το σκεφτεί λοιπόν η Επιτροπή. Μας ευχαριστώ. Κυρία Λόβεν. Ευχαριστώ. Βασικά έχω Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, γιατί πράγματι είναι δύσκολο να προσπαθεί κανείς να κάνει την ευθυγράμμιση και επίσης ε, την τροποποίηση και να μην τα μπλέξει και αυτά τα δύο. Αν συζητήσουμε μόνο την ε, λισαβονοποίηση, αυτό θα συζητήσουμε ή ε, και τα δύο. Colleagues have in their responses πριν περάσουμε σε δύο συζητήσεις για την έκθεση δηλαδή, να ακούσουμε πρώτα απ' όλα τα περί της διαδικασίας ευθυγράμμισης και λησαβονοποίησης. Και εγώ με τα χαράς θα επανέλθω στο, στην ουσία μετά. Για τις ε, τροπολογίες για την έκθεση αυτή. Κύριε Λόβιν. Εγώ έχω καταλάβει ότι ο πρόεδρος μας είπε να τα πούμε ε, όλα μαζί. Εγώ ουσιαστικά για, την, για τις ουσιαστικές τροπολογίες είχα κάποιες ερωτήσεις. Ε, σε ό,τι αφορά όμως το θέμα της λισαβονοποίησης. νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο σχήματο και σας στηρίζουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, πραγματικά γίνονται προτάσεις που τροποποιούν σημαντικά την πρόταση της Κομισιόν, όπως είναι η τροπολογία 3. Επιστημονική Συμβουλή μείωση κατά 25% προτείνει κομισιόν ή άλλα μέτρα. Και η ΣΥΤΡΕ στην πρότασή της λέει τα τάκ να ορίζονται μόνο για τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν κάποια α, απογεύματα όπως το Κάντεγα ο Γάδος που είναι σχεδόν στα πρόθερα της εξάλληψης. Σε σχέση με τη δεκαετία του 70 έχει μείνει το 1 ή το 2% του πληθυσμού αυτού. Και ότι αλλιεύεται, αλλιεύεται ως παρεμπίπτον αλλιεύμα, αλλά δεν είναι αποδεκτό αυτό λάβοντα υπόψη την κατάσταση του αποθέματος. και την με εξαφάνιση. Άρα εδώ διαφοροποιείται η απόψή μου σε σχέση με αυτήν της εισηγήτριας. Επίσης θα ήθελα κάποιες ε, επεξηγήσεις σε σχέση με την τροπολογία 5 όπου προτείνεται ως ώρα από την Κομισιόν τα 300 μέτρα. Βάθος δηλαδή μεγαλύτερο των 300 μέτρων και εσείς έχετε μια άλλη πρόταση. Δεν την έχετε βέβαια εξηγήσει ακόμη. Απλά σας θέτω το ερώτημα γιατί κάνετε αυτή την αλλαγή. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου, αφού η κυρία Τότσι που θα τα εξηγήσει όταν ξαναπάρει το λόγο αργότερα. Ευχαριστώ. Κυρία Φράγκα, η ερώτησή μου έχει να κάνει με τα σχέδια, με τα προγράμματα. Δεν έχω ε, κάποια ερώτηση προς την κυρία Ντότς. Θα ήθελα να μου απαντήσει ο κύριος Στίβενσον. Για να καταλάβουμε και να συμφωνήσουμε. Εγώ ξέρω ότι το Συμβούλιο η μειοψηφία αυτή που μπλοκάρει αυτά τα σχέδια αυτό που δεν θέλω σε καμιά περίπτωση είναι το Κοινοβούλιο να μπορεί να έχει λόγο σε ό,τι αφορά το Harvest Control Rule που κανονίζει το κατώτατο όριο και το ανώτατο όριο. Μέσα ε, σε αυτό το πλαίσιο μπορεί κανείς να κινηθεί. Έχουμε τη σημότητα και, τα παρά, και άλλες παραμέτρους σημαντικές. Όλα αυτά είναι τα κριτήρια για την καθιέρωση των ΤΑΚ. Εμείς εδώ στο Συμβούλιο Είπαμε ότι μεταξύ του ανώτατου και κατώτατου δεν θα τοποθετηθούμε. Το προσφέραμε αυτό στο Συμβούλιο. Αυτή είναι η μέγιστη δυνατή ευελιξία και η καλύτερη προσφορά μας προς το Συμβούλιο. Όμως, το Harvest Control Rule, να το ε, βγάλουμε εντελώ από την ε, συναπόφαση, ισοδυναμεί με το να αφήσουμε στα χέρια του Συμβουλίου την πλήρη ε, διακριτική ευχέρεια να καταρτίζει τα ΤΑΚ. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Επίσης, ο ίδιος ο κανονισμός, ο βασικός κανονισμός απαγορεύει στο να δοθεί στο Συμβούλιο εξουσία αυτή. Τι θέλει το Συμβούλιο λοιπόν. Πρώτα απ' όλα εμεί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μα. Συμφωνούμε να αφήσουμε την εξουσία αυτή στο Συμβούλιο, διότι αν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε στο Συμβούλιο την εξουσία, θα συμφωνήσει να πάμε στη συναπόφαση στο Συμβούλιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σα το λέω αυτό προκαταβολικά. Εγώ όμω δεν συμφωνώ με αυτή την απόφαση. Αν όμω οι περισσότεροι συμφωνούν, α προχωρήσουμε και θα έχουμε λύσει και το πρόβλημα. Το πρόβλημα, και νομίζω τον γνώρισε και το είπα τέλο πάντων μπροστά και στην Επίτροπο πριν, είναι με τον κανόνα αυτόν, το Harvest Control Rule. Θέλουμε να αφήσουμε ε, τελείω ελεύθερο το συμβόλαιο να κάνει ό,τι θέλει με τα ΤΑΚ. Θέλουμε να είναι καθαρά πολιτικό το θέμα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Κυρία Ντότς, παρακαλώ. Κοιτάξτε, ε, θα ήθελα να επανέλθω σε ορισμένα θέματα. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση του κυρίου Στίβενσεν ε, και νομίζω θα συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι στην Επιτροπή. Ε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή τη μεξικανική συμφωνία. Δεν είναι προς όφελος της βιώσιμης αλίας, ούτε του τομέα, ούτε της ε, πολιτικής ε, κατεύθυνσης ε, που πρέπει να χαράξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή μας έχουν στείλει εδώ για να κάνουμε ορισμένα πράγματα και αυτά πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος ε, μηχανισμός ε, για να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό. Ε, με την Ιρλανδική Προεδρία υπάρχει μια αχτίδα φωτός και μέχρι τώρα νιώθω απογοτευμένη γιατί δεν έχουν προάγει αυτό που θα μπορούσε να αποτελεί συμβιβασμό σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, δεν πιστεύω ότι τελικά θα περάσουν όλοι το δικό τους. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει κάποιος ε, μηχανισμός ε, για να λειτουργήσουμε. Στις ε, τροπολογίες που έχω συμπεριλάβει στην έκθεση προσαρμογής, εκεί δεν δίνω το πράσινο φως στο Συμβούλιο, Θεωρώ ότι πρέπει να ακούσουμε την άποψη της Επιστημονικής Επιτροπής επί του θέματος. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πρέπει να αναζητήσουμε ένα τρόπο για να προχωρήσουμε και ίσως τελικά να καταλήξουμε στο δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να επωφεληθούμε από την αχτίδα φωτός που προσφέρει η Ιρλανδική Προεδρία. Θα ήθελα να συζητήσω μαζί τους όταν θα έχουμε καταλέξει στην πρότασή μας, αλλά σε όσους παρίστανται εδώ σήμερα από την Προεδρία, θέλω να τους πω ότι αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο επιθυμούμε να αναβάλουμε συνεχώς. Όλοι ανησυχούν για το θέμα δεν μπορούμε να δρανίσουμε, ε, γιατί αυτό ίσως ε, να αρέσει το Συμβούλιο, αλλά εμείς θέλουμε να το λύσουμε το θέμα. Και δεν νομίζω ότι ε, το να καταφύγουμε σε δικαστήρια αυτή είναι η λύση του θέματος. Έτσι κι αλλιώς έχουμε ήδη καθυστερήσει επ' αυτού για δύο ολόκληρα χρόνια. Και επιτρέψτε μου να επανέλθω σε μια πιο ουσιαστική έκθεση που κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντική Ευχαριστώ λοιπόν τους ε, συναδέλφους για τα σχόλια τα οποία έχουν κάνει. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Σε αντίθεση με αυτά που συνέβησαν το Δεκέμβρη, πρέπει να προετοιμαστούμε για το μέλλον των αποθεμάτων γάδου. Νομίζω λοιπόν εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε στην Επιτροπή μας είναι το εξής. Κατά την άποψή μου, η τροποποίηση αυτή στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ε, γάδου είναι ένα ενδιάμεσο μέτρο. Και αυτό ε, θα πρέπει να την καταστήσουμε με ένα πρόγραμμα πολλών ειδών. Αυτό λοιπόν που προσπαθώ να κάνω είναι να προσφέρω κάποια ε, κάποιο ξεκαθάρισμα, αλλά πάνω απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε την αρχή ότι τα ε, επιστημονική φύσεως θέματα είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να λαμβάνονται διαρκώς υπόψη. Πρόσφατα ακούσαμε σχόλια από την Επιστημονική Επιτροπή και ακούσαμε ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια όπου υπήρξαν προσπάθειες να αυξηθεί ο πληθυσμός. Ε, πλέον ε, διαπιστώνεται μία μείωση των αποθεμάτων. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας ε, που πρέπει να γίνει. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και ο στόχος των τροπολογιών είναι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση εκείνη, την κατάσταση ε, σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής ε, και την τροποποίηση του προγράμματος του 2008. Η Ιζαμπέλα εξέτασε την ε, τροπολογία 3 που θεωρεί ότι μπορεί να τη στηρίξει και εγώ προσβλέπω στο να υπάρξει μια συζήτηση σχετικά με αυτές τις τροπολογίες για να δούμε κατά πόσον πράγματι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστική πρόταση σε προτάσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση που υπάρχει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα υπάρξει αυτή η συζήτηση. Είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό για την Επιτροπή μας να καταλήξουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό συμφωνίας σχετικά με την έκθεση. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα καθοριστικό μήνυμα που θα εκπέμψουμε προς το Συμβούλιο σχετικά με την έκθεση αυτή. Έτσι λοιπόν προσβλέπω στο να υπάρξει μια περαιτέρω συζήτηση μαζί σας επί του θέματος. Επίσης, προσπάθησα στις τροπολογίες μου να επεκτείνω τη συνεργασία ανάμεσα στον κλάδο και τους επιστήμονες. Ε, μέχρι τώρα όμως υπήρξαν πάρα πολλά εμπόδια και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εγώ προσπάθησα ε, οι συμβουλές ε, σχετικά με τη μείωση των ε, απορρίψεων. Νομίζω αυτό βολεύει όλους, όλοι θα κερδίσουν από αυτό και προς, εκεί, προς εκεί πρέπει να κατευθυνθούμε. Τροπολογία 6. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική τροπολογία. Ο εξοπλισμός που έχει περάσει μέσα από την διαδικασία των, της σταδιακής ε, εξέλιξης, τα κράτη-μέλη ίσως θεωρήσουν ότι είναι λογικό, εφόσον το έχουν πράξει αυτό και το έχουν βιώσει, να το επεκτείνουν ε, και, στα, και σε άλλα κράτη-μέλη. Επιπλέον, Ορισμένα κράτη-μέλη ε, έχουν προσαρμόσει καλύτερα τον κανονισμό. Ίσως ε, λοιπόν ε, πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω και το θέμα αυτό. Κατά τα άλλα, ορισμένοι αναφέρονται στις ροπολογίες 8 και 9. Εγώ νομίζω τα προγράμματα αυτά ε, αποδείχθηκαν επιτυχημένα και αυτή είναι μια πρωτοβουλία που πρέπει να την ενθαρρύνουμε, πρέπει να ε, προσπαθήσουμε ε, να διαδοθεί περαιτέρω αυτή η τροπολογία. Τώρα, αυτή η τροπολογία 9 σχετικά με το βάθος των 300 μέτρων. Η Επιτροπή δεν μας εξήγησε γιατί κατέληξε στα 300 μέτρα. Βεβαίως ε, έχω καταλάβει ότι ορισμένα κράτη-μέλη ε, διαφωνούν από αυτού και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ελέγξουμε εντελεχέστερα. Συνάδελφοι, αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη δουλειά και επίσης ε, επίμαχη Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε πολύ καλές τροπολογίες ε, επί του ε, προγράμματος 2008 έτσι ώστε να προσφέρουμε μεγαλύτερη σαφήνεια. Είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή αυτή να καταλήξει με συνένεση σε μία άποψη που θα μπορεί να την καταθέσει στο Συμβούλιο. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα σημαντικό μήνυμα προς το Συμβούλιο, ότι η Επιτροπή μας είναι ενωμένη και προσπαθεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα. Προσβλέπω λοιπόν σε περαιτέρω συζητήσεις σε μεσάς επί του θέματος. Ε, περιμένω τις ε, τροπολογίες σας. Ε, ο στόχος είναι να επιτύχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια, να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη αλία, τα βιώσιμα αποθέματα. Και νομίζω ότι επ' Ε, μπορούμε όλοι να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε το στόχο μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος το λόγο από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις δύο εκθέσεις. Σε δύσκολες συνθήκες. Δεν θα μιλήσω για το διαθεσμικό διέξοδο στο ζήτημα του πολιτού προγραμματισμού. Το κάνατε, σας τα είπε και η Επίτροπος. Υπογραμμίζω απλά ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει αν θα πάει ή όχι στο δικαστήριο, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε την απόφαση του δικαστήριου. Πρέπει να υπάρξει πρόοδος ούτως ή άλλως και να βρούμε έναν καλό τρόπο θεσμικής επίλυσης του θέματος. Δεν θα κάνω άλλα σχόλια. Για τις τεχνικές τροπολογίες τώρα. Δεν μπορώ να πω σε πολλές λεπτομέρειες για τα τεχνικά θέματα. Ίσως επειδή είναι να είναι απλούστερο να προχωρήσουμε σε μία τεχνικού διμερούς χαρακτήρα ανάλυση ε, εξηγώντα τις προτάσεις μας. Προφανώς η Επιτροπή ήθελε να απλοποιήσει όσο περισσότερο γίνεται τον υφιστάμενο κανονισμό. Κάποιες αλλαγές που προτείνουμε είναι τεχνικές, αλλά βασίζονται στην ε, τις συζητήσεις που είχαμε στο παρελθόν με τον κλάδο. Η πρότασή μας προσπαθούσε να απλοποιήσει. Κάποιες από τις τροπολογίες νομίζουμε, αλλά μπορεί να είναι θέμα διευκρίνησης, κάποιες έλεγα κάνουν λίγο πιο περίπλοκη τη διαδικασία. Δεν θα μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Επαναλαμβάνω ότι ίσως ήταν σκόπιμο να έχουμε μια τεχνικού χαρακτήρα συζήτηση με την κυρία Ντότ για να καταλάβουμε τα τεχνικά θέματα. Πάντως ο στόχος μας είναι να δώσουμε μεγαλύτερη διαφα... σαφήνεια και να επιτρέψουμε βιώσιμες... βιώσιμη αλληλεία και βιωσιμότητα του αποθέματος. Προς, τα... Προς εκείνη την κατεύθυνση δουλεύουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλετε ξανά το λόγο, κυρία Ντότζ. Um, that's, I'm happy, content to leave it, um, and uh, my door is open. Όχι. Ε, περιμένω τα σχόλια της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε. Ωραία, ολοκληρώθηκε και η συζήτηση. Προθεσμία για την υποβολή των απολογιών είναι η 25η Φεβρουαρίου. 12 το μεσημέρι. 25 του μηνός 12. Πριν κλείσουμε το θέμα αυτό, με ρώτησε ο Αντιπρόεδρος αν η νομική υπηρεσία μπορούσε να, μπορούσε να μας δώσει, να μας κάνει μια παρουσίαση, ανάλυση, εξήγηση για την ε, υπόθεση που ανέφερε η κυρία Δαμανάκη και το και η κυρία Ντόντ. Μπορούν να μας πούν κάτι. Θέλετε να ανοίξουμε μια παρένθεση και να δώσω το λόγο στην νομική υπηρεσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνει το λόγο. Πρόκειται για μια πολύ κρίσιμη στιγμή σεβασμού της συνθήκης της Λισαβόνας ο, η υπόθεση αυτή για την οποία είναι η συγγήτρια η κυρία Ντότς εντάσσεται πλήρως στο σημείο αυτό. Ήδη είχαμε σαφή μηνύματα από το Συμβούλιο για το τι θα κάνει και το τι έχει ήδη κάνει. Στις 19 12 με, κανονισ... με τον κανονισμό 1243 του 2012 το Συμβούλιο ενέκρινε μονομερός με τη νομική βάση του άρθρου 43.3 ιδία πρωτοβουλία διατάξεις που περιλαμβάνονταν στην πρόταση της Επιτροπής για τις προσαρμογές του πολιετούς ε, ε, προγράμματος ε, γάδου για τα 9, που περιέχονται στο άρθρο 9 και 12 του κανονισμού και είναι αντικείμενο των τροπολογιών 3 και 10 στην έκθεση. Έχουμε λοιπόν την κατάσταση ότι αυτή τη στιγμή ισχύει ήδη μία νομική πράξη αμφιλεγόμενης νομιμότητας, αλλά νομική πράξη παρατάφτα που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο. Ήδη λοιπόν είναι εφαρμοστέα νομοθεσία στην Ένωση, τα άρθρα 9-12 όπως τροποποιήθηκαν από τον κανονισμό που προανέφερα. Νομικά λοιπόν, με αυστηρά νομική ε, διάσταση, δεν έχουμε πλέον περιθώριο διαπραγμάτευση. Η μόνη λύση για να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας και να έχουμε ένα δικαίωμα λόγου ως προς το πώς υπολογίζονται τα τάκ σε μια περίπτωση όπου δεν είναι επαρκή η επιστημονική συμβουλή ή τι αυτοματισμός χρειάζεται, πρέπει να πάμε στο δικαστήριο γιατί το Συμβούλιο ήδη υιοθέτησε ένα νομικό κείμενο και δεν μπορεί καν να διαπραγματευτεί πλέον. Η μόνη λύση είναι το δικαστήριο. Και το μόνο που το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει είναι, το, το Κοινοβούλιο το μόνο που μπορεί να αποφασίσει είναι ότι να ζητήσει, να πείτε ότι ο πρόεδρος του θεσμικού οργάνου αποφάσισε μετά από διαβούλευση της νομικής επιτροπής να ζητήσει από την νομική υπηρεσία να προχωρήσει σε, στην εξέταση παραπομπής του Συμβουλίου στο δικαστήριο για την έγκριση αυτών των δύο διατάξεων της ε, Επιτροπής. Αυτό που κάνουμε είναι να ετοιμάσουμε την προσφυγή μας που θα υποβληθεί το αργότερο 15 Μαρτίου. Από ό,τι γνωρίζω από την ε, νομική υπηρεσία της Επιτροπής το ίδιο πράγμα κάνουν και αυτοί. Θα είναι μια κοινή προσφυγή των δύο θεσμικών οργάνων. Αυτό είπε και η κυρία Ραμανάκη. Το επιβεβαίωσε δηλαδή. Ότι και η νομική υπηρεσία αυτό εξετάζει. Συνοπτικά, είμαστε ενώπιον ενό τετελεσμένου γεγονότος. Υπάρχει μία υιοθετημένη νομική πράξη που μας αγνοεί παντελώ. Αν θέλουμε να μιλήσουμε, να έχουμε λόγο και να μας σέβεται το Συμβούλιο στο μέλλον, η μόνη εναλλακτική είναι να πάμε τώρα στο δικαστήριο. Αν δεν μας νοιάζει αυτό, να μας... Να μην μας αφήνουν να πούμε κάτι, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε νομικά, ωστόσο, αν θέλετε να γίνει σεβαστή η συνθήκη, σας λέω το εξή. Υπάρχει ήδη απόφαση, θα πρέπει να υπάρξει απόφαση του θεσμικού οργάνου να πάει σε δικαστήρια. Τώρα για την προηγούμενη, για την τρέχουσα υπόθεση που ζήτησε να μάθει ο κύριος Στίβενς, πρόκειται για μια κοινή προσφυγή των δύο οργάνων, ημών και της Επιτροπής. Πρώτα ήμασταν εμείς και μετά ήρθε και η Κομισιόν τον προηγούμενο Φεβρουάριο-Μάρτιο κατά μια μονομερούς απόφαση του Συμβουλίου και πάλι που αποφάσιζε την μελλοντική πρόσβαση σκαφών Βενεζουέλας στα νερά της Γαλλικής Γουιάνας που κατά άποψή μας ήταν διεθνή συμφωνία και την άποψη αυτή και η Επιτροπή δηλαδή. Η Επιτροπή, της, η Επιτροπή την πρόταση έχει, την είχε υποβάλει με πρόταση για να λάβει την σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου και μετά μονομερός πάλι το Συμβούλιο άλλαξε το, εργαλείο, το νομικό εργαλείο, ε, τη νομική βάση, χρησιμοποιώντας ένα, μια νομική βάση την οποία εμείς μόνο γνώμη δίνουμε, όχι σύμφωνη γνώμη. Δεν δώσαμε γνώμη, αλλά το Συμβούλιο χωρίς την γνώμη του Κοινοβουλίου και πάλι με βάση το 43.3 και χωρίς τη συνένεσή μας ε, πήρε απόφαση. Αυτό είναι εξωτερική διάσταση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής, δεν είναι τα πολιετή προγράμματα, αλλά έχει να κάνει και πάλι την εφαρμογή του, με την εφαρμογή του F43. Το κατά πόσο δηλαδή το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει λέγειν. Στη συγκεκριμένο πλαίσιο στην σύμφωνη γνώμη ή όχι, για να μπορέσει η Ένωση να αναλάβει διεθνείς ε, ε, υποχρεώσεις στον τομέα της αλίας. Είναι δηλαδή το ίδιο άρθρο της συνθήκης σε άλλο πλαίσιο. Στους δύο αυτούς ε, εμείς προσφύγαμε κατά του Συμβουλίου για την ιστορία αυτή με τους Βενεζουελανούς. Για την τωρινή περίπτωση θα πρέπει να περιμένουμε τις οδηγίες από τον πρόεδρο Σούλτς. Οι δύο προσφυγές νομίζω ότι θα συμπληρώσουν με χρήσιμο τρόπο η μία την άλλη για να έχουμε και μία καθοδήγηση από το δικαστήριο. Μία τελευταία παρατήρηση, πρόεδρε. I Ως δικηγόρος δεν νομίζω ότι μπαίνουμε, πέφτουμε σε παγίδα, ακόμα και αν πάμε στο δικαστήριο. Διότι, επανελαμβάνω, ότι ήδη το Συμβούλιο έλαβε απόφαση, μονομερός, αποφάσισε. Δεν έχουμε δηλαδή νομικό κενό. Βεβαίω να έχετε πολιτικέ διαπραγματεύσει. Τίποτα δεν υποδείζει κάτι τέτοιο. Και προφανώ είναι κάτι θετικό. Προφανώ κάποια στιγμή πρέπει να ζητήσουν την άποψη του δικαστηρίου. Και αυτό δεν εμποδίζει το να έχουμε πολιτικές διαπραγματεύσεις. Αυτό ή σε άλλα πλαίσια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ντότς σε το λόγο και η κυρία Λόβιν. Κυρία Ντότς πρώτα. Ευχαριστώ. Αυτό που μας είπε ο συνάδελφος σίγουρα αποτελεί την ερμηνεία ενός νομομαθούς, αλλά πρόκειται για πολιτικά θεσμικά όργανα, άρα πρέπει να υπάρξει και ένα πολιτικό μονοπάτι, ε, στο πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να κάνουν τις πραγματεύσεις μας. Μπορεί πράγματι να συμβαδίζει ε, και αυτή η προσέγγιση, δηλαδή μια νομική ενδεχομένως δράση και μια πολιτική διαπραγμάτευση να πηγαίνουν εκ παραλίλου τα δύο αυτά. Εξακολουθώ πάντως να πιστεύω ότι θα πρέπει η Ιρλανδική Προεδρία να έχει κάποιο χρόνο στη διάθεσή της ε, ώστε να υποβάλει μια πρόταση που θα άρει αυτό το αδιέξοδο. Εγώ έχω μιλήσει με προσώπους άλλων κρατών μελών, όχι της δικής μου χώρας και ε, θα ε, χαίρονταν το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο μάλλον, η Κομισιόν να καταφύγουν στο δικαστήριο, γιατί αυτό θα παγώσει οποιαδήποτε πολιτική διαδικασία και διεργασία. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν να μου πείτε τι ακριβώς θα συμβεί μέχρι τις 15 Μαρτίου. Κυρία Λόβιν. Ήθελα να κάνω ένα πολύ έτσι πρακτικό ερώτημα. Νομίζω ότι οι δύο λύσεις αυτές που προτείνεται να ακολουθήσουμε είναι η σωστή προσέγγιση. Το πρακτικό μου ερώτημα είναι το εξής. Εάν ε, δρομολογήσουμε μία νομική διαδικασία ενώπιν του δικαστήριου, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή. Yes, Mr. President, of course. Θα μπορούσε να διακοπεί αυτή η διαδικασία. Ναι, βεβαίως μπορεί να διακοπεί αργότερα, είναι απάντη. Υπάρχει όμως ένα μια προθεσμία. 15 Μαρτίου είναι αυτή η προθεσμία. Μέχρι τότε δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε αν θα εμείνουμε σε εντολές που έχουμε, ε, έχουμε συμφωνήσει και αν θα προσφύγουμε στο δικαστήριο. Και αφού γύρουμε αυτή την αγωγή, φυσικά μπορούμε να την ε, καταλήψουμε ε, αφού λάβουμε βέβαια τη σχετική πολιτική απόφαση. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, κάποιες φορές ε, εκπλήσωμαι, γιατί νομίζω ορισμένες φορές ότι συμφωνούμε κάποια πράγματα και τελικά δεν τα κάνουμε. Έχουμε τις δύο επιλογές είτε να κάνουμε αυτά τα δύο, είτε να συνεχίσουμε την πολιτική διαδικασία. Φυσικά και μας έδωσε τη νομική της ερμηνεία υπηρεσία αυτή, η νομική μας υπηρεσία, αλλά μην τρελαθούμε, πρέπει να ε, δούμε τι θα κάνουμε τελικά. Στην τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών αποφασίσαμε ότι θα εξετάσουμε όλες τις απόφασεις οι οποίες παραβιάζουν την αρχή αυτή και όχι μόνο σε σχέση με όσες είχαν εγκριθεί τότε. Αυτό ήταν ε, αυτό που αποφασίσαμε νομίζω. και νομίζω ότι επικυρώνεται η διαδικασία που έχει επιλέξει το Κοινοβούλιο και με αυτά που μας πει νομική υπηρεσία. Δηλαδή κάνουμε ε, και συνεχίζουμε τις προσπάθειες στο πλαίσιο της πολιτικής διαπραγμάτευσης. Ε, αποδεσμεύσαμε τη διαδικασία για την έγκριση τελικά της έκθεσης Γκάλαχερ, αλλά πρέπει να καταφέρουμε στο δικαστήριο. Αυτή είναι η άλλη οδός. Παράλληλες είναι οι οδοί. Δεν ξέρω γιατί θα έπρεπε να τέμνονται κάπου. θα δούμε τι αποτέλεσμα θα προκύψει. Νομίζω ότι είναι σαφής ε, ο συλλογισμός μας ε, και το σκεπτικό μας. Δεν ξέρω, ε, νομίζω αυτό είχαμε συμφωνήσει. Ας πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της Μέση Διάθεσης, που είναι το τελευταίο για σήμερα, το πρωί. Α, κάτι ξέχασα. Για τις δύο εκθέσεις της κυρίας Ντότς, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. 25 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, 18 προς γενετικού τρόπου πόρου συγγνώμη, και δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή στα ωφέλη που προκύπτουν από την χρησιμοποίησή τους στην Ένωση. Ο κ. Χάτσον που δεν είναι εδώ, δεν τον βλέπω, θα ακούσουμε όμως ε, την ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α, η κ. Λόβιν μου ζητά Θα εκπροσωπήσετε τον κύριο Χάτσον. Λέβιν. Ναι, ήθελα απλά να σας πω ότι ο κύριος Χάτσον ζήτησε ε, συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, αλλά μου έδωσε κάποια ε, με κάποιες ερωτήσεις του. Ωραία. Να δώσουμε όμως πρώτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση που έχετε μπροστά σας ε, για κανονισμό έχει ως στόχο να εφαρμοστεί σε νοσιακό επίπεδο ένα πρωτόκολλο για την ε, βιολογική βιοπικιλότητα, ε, το πρωτόκολλο Ναγκόγια, επειδή ήταν αντικείμενο διαπραγματεύσεων στην Ιαπωνία. Εκεί προβλέπεται μια δίκαιη κατανομή των ωφελών που προκύπτουν από την εκμετάλλευση. Αυτό λοιπόν το στοιχείο της ισότιμης ε, κατανομής ε, είναι ένα, ένας από τους τρεις πυλώνες της ε, οικολογικής βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν συνυπογράψει αυτή τη συμφωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο Ναγκόγια που εξετάζει την πολιτική δέσμευση για ταχεία εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλου. Από την άλλη πλευρά, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν καλέσει επανειλημμένα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μέτρα ε, για την εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάστηκαν λοιπόν τον Οκτώβρη ε, του 2012 συγκεκριμένα μέτρα. Αυτή η πρόταση κανονισμού είναι το αποτέλεσμα μιας ευρείας διαδικασίας διαπραγματεύσεων. Διαπραγματευτήκαμε με εμπλεκόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε διμερείς επαφές ε, με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ε, εργαστήρια, σεμινάρια και επίσης ε, εκπονήσαμε και μία μελέτη αντικτύπου. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τομεακές μελέτες για να υπάρξει μία θέση για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με βάση αυτές τις πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοίμασε τη μελέτη αντικτύπου. Θα ήθελα λοιπόν να ε, προβάλλω κάποια χαρακτηριστικά αυτής της ε, κατευθυντήριας γραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται στη μελέτη αντικτύπου. Αυτή λοιπόν η μελέτη χρησιμεύσε ως ε, βάση για να κάνουμε τις συγκρίσεις μας σχετικά με τα καλύτερα δυνατά μέτρα. Τα βασικά λοιπόν χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Πρώτον, οι γενετικοί πόροι χρησιμοποιούνται για πάρα πολλούς στόχους από πολλούς παράγοντες που έχουν και διαφορετικά ε, συμφέροντα. Ε, διάφοροι παράγοντες παρεμβαίνουν σε διάφορες ε, φάσεις της αλυσίδας ασχολούνται με την έρευνα, τα προϊόντα και το καθεξής. Τρίτον, οι ε, μελλοντικές ε, έρευνες για τους γενετικούς πόρους ε, θα αυξηθούν ενώ η ζήτηση για πρόσβαση επιτόπου θα περιοριστεί στους περισσότερους τομείς. Τέταρτον, η χρήση παραδοσιακών γνώσεων σε συνδυασμό με τους γενετικούς πόρους ε, δεν μοιάζει να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και θα ε, περιοριστεί περαιτέρω. Πέμπτον, η in situ πρόσβαση κατά κύριο λόγο γίνεται από πανεπιστημιακούς ερευνητές και μελετητές ε, που σχετίζονται με έξεση του συλλογές. Κατόπιν έχουμε συλλογές έξεση του που καθορίζουν, καθοριστικό, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για ε, μη εμπορικούς και εμπορικούς χρήστες και τέλος ε, οι βέλτιστες πρακτικές αυτής της συνθήκης ε, υπάρχουν στην αλυσίδα χρηστών και δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο για τις δραστηριότητες downstream. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της συμφωνίας που έχει προκύψει από τη μελέτη αντικτύπου. Η μελέτη αντικτύπου βασίστηκε σε μία σειρά θεμάτων. Πρώτον, σε διάφορα μέτρα αναλύθηκαν αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της ε, προσπελασιμότητας ε, και ε, το θέμα του χρήστη. Το σημείο κίνησης που χρησιμοποίησαμε ήταν μέγες, της ευκαιρίας χρήσης των γενετικών πόρων. Αυτό σημαίνει ότι μεγιστοποιούμε ε, και την βιολογική ε, ποικιλομορφία. Τα βασικά κριτήρια που μας καθοδήγησαν στην προσέγγιση μας ήταν πρώτον η ε, συμμόρφωση Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πρωτόκολλο, δεύτερον η κατάργηση της νομικής ασφάλειας για τους χρήστες, κατόπιν να μπορεί να γίνει έρευνα, κατόπιν τέταρτον δηλαδή τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβαδίζουν με τις υπάρχουσες πρακτικές έκτον να λαμβάνει κανείς υπόψη του το κόστος ε, στην αλυσίδα της ε, των ερευνών και τέλος να επιμερίζεται το ε, διοικητικό κόστος. Με βάση όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καταρτήσαμε αυτήν την πρόταση κανονισμού. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας προβάλλω τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της ε, πρότασης. Υπάρχουν έξι βασικά στοιχεία στην πρόταση αυτή. Πρώτον, οι χρήστες ε, είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν ε, την απαραίτητη διδέουσα επιμέλεια. Κατόπιν να υπάρχει ένα δίκαιο σύστημα συλλογών, να αναγνωρίζονται οι βέλτιστες πρακτικές, να ελέγχεται η συμβατότητα των χρηστών, να υπάρχει μια πλατφόρμα και δυνατότητα πρόσβασης σε συζητήσεις, ανταλλαγές πληροφοριών και το καθεξής, έκτον να υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας κατά την εφαρμογή δηλαδή να υπάρχει μια βάση για περαιτέρω συνεργασία με τρίτες χώρες και άλλες περιοχές. Θα ήθελα λοιπόν να εστιάσω την προσοχή μου σε ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα. Πρώτα απ' όλα ε, στην υποχρέωση της δέουσας επιμέλειας. Αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό που διατρέχει τον κανονισμό. Με βάση λοιπόν αυτήν την υποχρέωση, όλοι οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια για να διασφαλίζουν ότι οι γενετικοί πόροι και οι γνώσεις σχετικά με αυτούς προσφέρονται με βάση τις ε, νομικές προϋποθέσεις που ισχύουν και με τον τρόπο αυτό τα ωφέλη που προκύπτουν επιμερίζονται δίκαια. Επιπλέον, όλοι οι χρήστες πρέπει να παραδίδουν στους επόμενους χρήστες τις πληροφορίες που είναι σημαντικές. Επιπλέον, οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να εξάγουν συμπεράσματα από όλες αυτές τις πληροφορίες, να διερωτώνται δηλαδή κατά πόσον ε, όλα αυτά είναι συμβατά με την κείμενη νομοθεσία. Και τέλος, εφόσον υπάρχει παραβίαση της ε, υποχρέωσης για την δέουσα επιμέλεια, αυτή η παραβίαση να συνεπάγεται κυρώσεις. Υπάρχει και μία άλλη πολύ σημαντική διάταξη που αφορά στην σύσταση ενός ε, ευρωπαϊκού ενωσιακού συστήματος ε, περί ε, συγκέντρωσης δεδομένων. Υπάρχουν φοβερά παράσιτα στο μικρόφωνο του μιλτή. Λυπάμαι πολύ. Αυτή λοιπόν η διάταξη σημαίνει ότι εάν υπάρχει η συγκέντρωση δεδομένων θα πρέπει όλα αυτά να συμβαδίζουν πλήρως με ε, δείγματα γενετικών πόρων. Επιπλέον, οι χρήστες ε, οι οποίοι θέλουν να έχουν γενετικούς πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια, κάτι που ισχύει κατά την αναζήτηση όλων των πληροφοριών. Και τέλος, το σύστημα της ε, ενωσιακής συγκέντρωσης δεδομένων ε, πρέπει να ωφελεί τους ακαδημαϊκούς ερευνητές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια δεύτερη σημαντική διάταξη του κανονισμού. Η τρίτη σημαντική διάταξη έχει σχέση με την αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ενώσεις χρηστών μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να αναγνωρίσει ένα συγκεκριμένο συνδυασμό διαδικασιών, εργαλειών και μηχανισμών που αναπτύσσει μια ένωση και αυτά να ε, χαρακτηριστούν ως βέλτιστη πρακτική. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι υποχρεωμένες ε, να λαμβάνουν υπόψη τους ότι αυτή η βέλτιστη πρακτική μειώνει τον κίνδυνο μη συμβατότητας του χρήστη και διευκολύνει και αιτιολογεί και τους ελέγχους. Και τέλος, η επίσημη αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών αυξάνει την νομική ασφάλεια, μειώνει το κόστος για τους χρήστες και για τη δημόσια διοίκηση. Πάμε τώρα στην τέταρτη βασική διάταξη του κανονισμού που είναι ο έλεγχος της ε, συμβατότητας των χρηστών και των σημείων ελέγχου. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν σε συγκεκριμένα σημεία ότι είναι συμβατοί ε, σχετικά με την δέουσα ε, επιμέλεια. Αυτά τα σημεία ελέγχου θα κρίνουν κατά πόσον οι χρήστες πράγματι τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Οποιαδήποτε παραβίαση του κανονισμού από τους χρήστες συνεπάγεται κυρώσεις ε, και αυτό με, ε, αποτελεσματικές, με αποτελεσματικό τρόπο. Θα ήθελα ή θέλησα να ε, προβάλλω αυτές τις τέσσερις βασικές διατάξεις του κανονισμού. Ο κανονισμός αυτός συζητιέται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο, ε, στην Επιτροπή και επίσης συζητιέται ο κανονισμός και στο Συμβούλιο. Και επίσης ε, έχουμε καταθέσει και μία πρόταση για επικύρωση του πρωτοκόλου της Ναγκόγια. Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε λοιπόν η Επιτροπή είναι στη διάθεσή σας των Ευρωβουλευτών για οποιαδήποτε διευκρίνηση επιθυμείτε. Ε, Ευχαριστώ κυρία Λοβέν. Ευχαριστώ. Όπως είπα, εξ ονόματος του κύριου Χάτστον, πρώτον, ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους, ζητεί συγγνώμη από τους συναδέλφους στην Επιτροπή, δεν μπορούσε να έρθει σήμερα, λόγω ανηλμένων υποχρεώσεων στη Σκοτία. Συγγνώμη, λέει. Θα σας διαβάσω τι μου γράψε. Καλωσορίζω την πρόταση της Επιτροπής που έχει στόχο να υλοποιήσει το πρωτόκολλο της Ναγκόγιας. Η Σύμβαση για την Βιολογική Επικοινότητα θέτει σημαντικές αρχές που αφορούν τα κυρίαρχα δικαιώματα στους γενετικούς πόρους μεταξύ των οποίων τα δικαιώματα των αυτόχθονων και τοπικών κοινοτήτων. Ωστόσο, δεν παρουσιάζει σαφώ πώς εφαρμόζονται τα δικαιώματα αυτά το πρωτόκολλο της Ναγκόγια και οι πρώτες επιτροπής προσπαθούν να καλύψουν το πρόβλημα αυτό. Η ουσία του πρωτοκόλλου δεν έχει επιπτώσει στη διαχείριση της ασέλειας στενή ταινία, ωστόσο το κείμενο ρητά αναφέρει μεταξύ των βασικών τομέων με τους οποίους ασχολείται είναι η διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας δεδομένου ότι η Επιτροπή μας ε, στις ευθύνες της έχει και την διατήρηση των αλληλευτικών πόρων, είναι ότι το πρωτόκολλο υπάγεται στον τομέα αρμοδιοτήτων ε, της Επιτροπής μας. Το πρωτόκολλο επιτρέπει στις αναπτυσσόμενες χώρες και τους αυτόχθονες πληθυσμούς να εκμεταλλευτούν καλύτερα τους ε, γενετικούς πόρους στους οποίους έχουν κυριαρχία. Ε, αυτό είναι βασικό ε, συμφέρον της χώρα, των λαών αυτών και είναι κρίσιμο λοιπόν το ότι προσπαθείτε σαν Επιτροπή να καλύψετε το κενό αυτό. Ο κύριος Χάτσον ήθελε μια σειρά διευκρινήσεων από πλευράς Επιτροπής στις εξής ερωτήσεις. Το άρθρο 13 του πρωτοκόλλου αναφέρει ότι κάθε χώρα θα ορίσει ένα ενιαίο ένα ενιαίο, ε, μια ενιαία ε, δομή, μια ενιαία αρχή. Το άρθρο 13 του πρωτοκόλου αναφέρει ότι κάθε πλευρά θα ορίσει μια ε, ενιαία δομή ως focal point με αρμοδιότητε σε εθνικό επίπεδο. Μπορεί επίσης να ορίσει μια, μια ξεκάθαρη, ξεχωριστή δομή για το σκοπό αυτό. Το άρθρο 6 της ε, τη επιτροπή αναφέρει ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει μία ή περισσότερες εθνικές αρχές και η Επιτροπή θα ορίσει ένα σημείο επαφής, focal point. Πρώτη ερώτηση. Αυτό σημαίνει ότι το σημείο επαφής της Επιτροπή θα είναι το μόνο και για τα 27, ένα δηλαδή, αντί των εθνικών σημείων επαφής ή τα εθνικά σημεία επαφής θα υπάρχουν και σε επίπεδο κάτω από αυτά της ενωσιακής, του ενωσιακού σημείου επαφή. Η δεύτερη ερώτηση αφορά στο ευρύτερο πλαίσιο της Σύμβασης για τη βιοποικιλότητα πώς ορίζονται τα ε, κυρίαρχα δικαιώματα βάση των ε, ενάλλειων πόρων ε, στα χωρικά ύδατα ή και στη, στα διεθνή ύδατα θα μπορούσε η Επιτροπή να κάνει αυτή τη διευκρι... να διευκρινίσει αυτά τα σημεία. Ευχαριστώ. Άλλος, θέλει το λόγο. Κομισιόν, θέλετε να απαντήσετε. Thank you, Mr. Chairman. With regard to the, the, the second question, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το δεύτερο θέμα, προφανώς η ευέλεια του κανονισμού είναι να καλύψει πόρους μέσα στη δικαιοδοσία των κρατών μελών της Ένωσης. Άρα η απάντηση είναι στα χωρικά ύδατα. Για τη δεύτερη ερώτηση ίσως είναι καλύτερα να απαντήσει συνάδελφός μου. Ευχαριστώ. Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια απαιτεί από κάθε συμβαλόμενο μέλος να ορίσει ένα σημείο επαφής το σημείο επαφής της Επιτροπής δεν υποκαθιστά το σημείο επαφής των κρατών μελών. Ορίζουν ένα σημείο επαφής καθώς και εφόσον εγκρίνουν το πρωτόκολλο δεν θα ήθελαν τα κράτη-μέλη να έχουν ένα μόνο σημείο επαφής, νομίζω. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Σας ευχαριστώ όλους. Θα ξεκινήσουμε στις 3 με την ακρόαση για τα είδη βαφέων υδάτων προς μια βιώσιμη αλληλεία. Ευχαριστώ και καλή σας όρεξη.